δελτίο και βέβαια όπως συνήθως ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και ο κύριος ε, Πίπερ έχει αποσυρθεί ως αναπληρωτής και το ΕΛΚ θα πρέπει να ορίσει τον αντικαταστάτη του. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις ε, της Προέδρου και τώρα πάμε στο σημείο 3. Έχουμε την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα ε, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα λεγόμενα hot spots σε Ιταλία και Ελλάδα. Έχουμε την κυρία Κίνικη και τον κύριο Ντεγιόν συνεισηγητές. Αλλά πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω. E σήμερα την ειδική έκθεση για τα hot spots, τα κέντρα υποδοχής ε, και ταυτοποίησης. Στο διάστημα του 2015 και 2016 το δικαστήριο αποφάσισε να προσεγγίσει το θέμα των hot spot. Εκτιμήσαμε την ε, λειτουργία αυτών των κέντρων στην Ιταλία και στην Ελλάδα από τη στιγμή που για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν το Μάιο του 2015 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2016. Επικεντρωθήκαμε σε δύο θέματα. Πρώτον, που βρισκόντουσαν τα κέντρα αυτά αν είχαν δημιουργηθεί εγκαίρως και αν είχαν τις απαραίτητες δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες με βάση ε, τις οδηγίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης. Και δεύτερον, αν ήταν αποτελεσματικά στη διαχείριση της ροής των μεταναστών, επιτρέποντας ε, την εγγραφή, την καταγραφή και την ε, ε, δακτυλοσκόπηση των μεταναστών. Το ερώτημα είναι αν πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και οι διάφοροι οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν. Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται, τότε το ε, σύστημα μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να κινδυνεύσει με κατάρρευση. Στη διάρκεια της προσέγγισης μας είδαμε ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα που τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο που ξεπερνά και όπου συνθήκες που ξεπερνούν τις δυνατότητες του κέντρου μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά του. Είναι σημαντικό να καταγράψουμε ότι δεν ελέγξαμε τις εθνικές διαδικασίες συνέχισης όσον αφορά το άσυλο. Το βασικό, το βασικό συμπέρασμά μας είναι ότι μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει η προσέγγιση των κέντρων ε, υποδοχής και ταυτοποίησης των hot spots στο σύστημα έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν στρατηγικό μέρος του σχεδίου για μια οργανωμένη ανταπόκριση σε μια ε, κατάσταση που ταχύτατα προχωρούσε προς ανθρωπιστική καταστροφή. Επιπλέον καταλήξαμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και γι' αυτό έχουμε κάνει πέντε συγκεκριμένες προτάσεις που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση της μετανάστευσης. Πρώτον, η ανάγκη να ανταποκριθούμε στην ανεπαρκή δυναμικότητα των hot spot, καταρχήν αναβαθμίζοντας τις υποδομές και στην περίπτωση της Ιταλίας να αυξηθεί ο αριθμός τους κατά δύο, όπως είχε αρχικά Επίση, προβλεφθεί. Επίσης συνιστούμε όλοι οι παράγοντες να κάνουν περισσότερα για να εξασφαλιστεί η επαρκής αντιμετώπιση του θέματος των ασυνόδευτων ανηλίκων. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι κατάλληλοι χώροι για αυτούς και να διεκπεραιώνεται γρήγορα η διαδικασία ασύλου. Επιπλέον επιμένουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να επιμείνει στον διορισμό ε, στελεχών για την προστασία των ε, ανηλίκων. Επίσης, Θέλουμε η Κομισιόν να συνεχίσει να επιμένει για την, στην χρησιμοποίηση αυξημένου αριθμού ειδικών ε, σε εθνικό επίπεδο με τις απαραίτητη τεχνογνωσία και την ε, ε, επαρκή διάρκεια της θητείας. Επιπλέον πρέπει η Κομισιόν να αξιολογήσει αυτή την προσέγγιση που είναι σημαντική για την επαρκή διαχείριση της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση που μας παρουσιάσατε. Οι δύο συνεισηγητές, ποιος θέλει να ξεκινήσει, ε, κυρία Κινίτσι. Παρακαλώ κύριε Κινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την παρουσίασή της έκθεσης. Πράγματι έφτιαξε πολύ σημαντικά στοιχεία του συστήματος των Χωστότ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο De για την εξαιρετική συνεργασία, για το έγγραφο εργασίας και για την συνεργασία και για το πνεύμα με το οποίο εργαστήκαμε επί του κειμένου. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, όπως ακούσαμε, μας δείχνει και ποια είναι τα κρίσιμα σημεία στην διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Η απάντηση της Ένωσης ε, δυστυχώς απέναντι στην κρίση αυτή ήταν ίσως ακατάλληλη και ενίοτε αναποτελεσματική στην πραγματικότητα άφησε τις ε, χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι στην πρώτη γραμμή μόνες τους η βοήθεια που είχε ενεργοποιηθεί και η υποστήριξη του ΕΑΖΟ, της Frontex και της Europol ε, υπήρξε παρόλα αυτά, ήταν ανεπαρκής για τη διαχείριση μιας συνεχούς μεταναστευτικής ροής. Αυτό οδήγησε την Ελλάδα και την Ιταλία να χρειαστεί να ε, χρησιμοποιήσουν επιπρόσθετους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να αντιμετωπίσουν αυτή την υποδοχή. Και οικονομικά αλλά και σε ανθρωπίνους πόρους χρειάστηκε να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις χώρες αυτές και όλη η προσπάθεια έπεσε στις ώμους των δύο αυτών χωρών. Αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, παραδείγματο χάρη, εγώ αναφέρομαι στα στοιχεία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευση. Η, από την αρχή του χρόνου έχουμε πάνω από 100.000 μετανάστες που έχουν περάσει την Μεσόγειο και το 80% έχουν φτάσει στην Ιταλία, 80.000 δηλαδή, και οι υπόλοιποι στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα των hot spot ε, στην πραγματικότητα λειτουργεί ε, και υπάρχουν ε, κάποιες ελλείψεις και κάποια προβλήματα, όπως μας είπε και το ηλεκτρικό συνέδριο. Έτσι λοιπόν, αν δούμε αυτή την κατάσταση της συνεχούς ροής ατόμων που φτάνουν στην επικρατειά μας και ιδίως στις ακτές της Σικελίας, της Ιταλίας γενικότερα και της Ελλάδας, πιστεύουμε ότι το Ταμείο Μετανάστευσης ε, ε, και στο Ταμείο Ασφάλειας θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι κανόνες για να χορηγηθούν έκτακτες βοήθειες, γιατί χρειάζεται γρηγορότερη αντίδραση απέναντι στις ανάγκες αυτές. Όμως, κυρίω πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι στι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να βελτιωθούν οι δομέ φιλοξενίας. Γιατί πρόκειται για μια δαπάνη η οποία δεν μπορεί να βαραίνει μόνο του εθνικούς προπολογισμού. Στην πραγματικότητα πρέπει να πούμε ότι αν και με τις δυσκολίες ε, με τις οποίες λειτουργούν τα hot spot, τουλάχιστον στην Ιταλία, το 100% των μεταναστών καταγράφεται τακτικά. Βλέπετε λοιπόν ότι δίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα αυτό στα hot spot. Και χαίρομαι που αναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ε, υπάρχει ειδικό προσωπικό που τους υποδέχεται υπάρχει και άλλη μια πτυχή που θέλαμε να θίξουμε, δηλαδή τον ε, κίνδυνο που διατρέχουν κυρίως οι ανήλικοι, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Βέβαια ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλός αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό χρειάζεται όχι μόνο να εμβαθύνουμε περαιτέρω, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται και μια πρόσθετη υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τα νομοθετικά μέσα και όχι μόνο Europol, Eurojust και Frontex εργάζονται για να υποστηρίξουν τις εθνικές αρχές για την καταπολέμηση των αδικημάτων αυτών που είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα. Όμως αντιμετωπίζουμε και δυσκολίες ε, ε, να αντιμετωπίσουν ε, τον αριθμό των μεταναστών οι οργανισμοί αυτοί καθώς δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν με το έγγραφο να καταδείξουμε ότι λειτουργούν τα hot spot. Ε, η Ιταλία εργάζεται για να ε, συμπληρώσει τον αριθμό των hot spot που προβλέπονται στη χώρα μου. Βέβαια, πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες στο θέμα αυτό. Και πάλι ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Ελευτικού Συνεδρίου και τον συνάδελφο Ντεγιόνγκ για την τεράστια συνεισφορά του για το έγγραφο εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφο De Jong, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ειδική αυτή έκθεση, τον κύριο Βέσπερκ. Πράγματι, συνεργάστηκα με πολύ μεγάλη χαρά με την κυρία Κινίτση για το έγγραφο αυτό εργασίας και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα δικά της λόγια για την συνεργασία μας. Νομίζω ότι και οι δύο αντιμετωπίσαμε ένα κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ειδική έκθεση. Και θεωρώ ότι συμφωνεί και το ελεγκτικό συνεδρίο ότι δηλαδή ουσιαστικά απεικονίζει ε, φωτογραφικά μια συγκεκριμένη ad hoc κατάσταση. Τα κέντρα αυτά ε, υποτίθεται ότι θα καταχωρίζουν τις αιτήσει ε, και θα ταυτοποιούν τους, ε, τους αφικνόμενους. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, υπάρχουν εξετάσεις των αιτήσεων, υπάρχουν ε, οι απορρίψεις και τι θα γίνει με την επιστροφή ε, των αιτούντων άσυλο. Πρέπει να δούμε δηλαδή την όλη αλυσίδα. Αν η όλη αλυσίδα δεν λειτουργεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι βιώσιμα αυτά τα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση, ιδίω λαμβάνοντα υπόψη του αριθμού. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλε αφήξει και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα. Αυξάνονται τα νούμερα πρόσφατα από ό,τι μου λένε οι Έλληνες συνάδελφοι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αλυσίδα, τελικά αυτά τα κέντρα δεν μπορούν να αποτελέσουν τη λύση από μόνα τους. Και αυτό ήταν και το πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με αυτή την ειδική έκθεση. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να είχαμε μια ευρύτερη, μια πλήρη εικόνα. Αν δείτε και την μεταγκατάσταση θα ε, καταλάβετε κι εσείς ότι δεν λειτουργεί όπως είχε προβλεφθεί κάποιες μετακαταστάσεις αλλά όχι στο βαθμό που είχε συμφωνηθεί στο παρελθόν. Και βέβαια αυτό προκαλεί συμφορήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις επιστροφές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί μια ευρωπαϊκή και αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Γιατί χρειάζονται προσπάθειες και με τις τρίτες χώρες, ε, να δεχθούν δηλαδή αυτές τις τρίτες χώρες τους επικόστου όταν αυτοί πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής. Το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και επιπροσθέτως, ε, στα όσα είπε η κυρία Κίνητση για κάποιες αναλυτικές πτυχές ε, που έχουν να τα απορίσματα της έκθεσης, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια ε, ένα follow-up. Θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την ειδική έκθεση. Βέβαια γνωρίζω ότι όλες οι ειδικές εκθέσεις του Ενεκτικού Συνεδρίου έχουν ε, τη συνέχεια ε, κάποια στιγμή, αλλά θα ήταν σημαντικό αυτό το follow-up να λάβει υπόψη όλη την αλυσίδα. Και έστω την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία επιστροφής εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο με αυτή την προσθήκη. Κατά τα λοιπά συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε η κυρία Κινίτσι για τα σημαντικά αυτά ε, σημεία. Ε, για τα παιδιά τα είπε πολύ καλά ε, και το ελληνικτικό συνέδριο τα τόνισε αυτά. Δεν βοηθάει επίσης το να φέρνει σε περιστασιακά. Χρειάζεται συνεχής παρουσία των εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να βοηθήσουν και νομίζω ότι το λέει και το Ελεκτικό Σύνδρο στα πορίσματά του. Αυτά από πλευρά μου και περιμένω βέβαια να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Η ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι απογοητεύτηκα με αυτήν την ειδική έκθεση. Ουσιαστικά δεν πρόκειται ούτε για ειδική έκθεση, ούτε για audit, ούτε για λογιστικό έλεγχο. Ουσιαστικά έχουμε μία περιγραφή των ε, διαδικασιών, αλλά δεν, ε, ξέρουμε τι γίνεται με τα χρήματα αυτά, με τα κονδύλια, δεν ξέρουμε αν επαρκούν ή όχι. Ε, έψαξα αλλά ματέως για να βρω κάτι σχετικό. Δεν έχουμε μια γενική εικόνα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, που και να μην είναι καν διαθέσιμα. Ε, το θέμα είναι όμως τι κάνουμε με αυτή την περιγραφή της κατάστασης και πώς απαντάμε στο ερώτημα αυτό για τους εμπειρογνώμονες για τη διάρκεια της παρουσίας και της εργασίας τους επιτόπου. Υπάρχει ε, κάποια δυνατότητα οι εμπειρογνώμονε που έρχονται και από τι χώρε από τι οποίε προέρχονται να αντιμετωπίσουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα να, εξειδικευμένα. Η συνάδελφο τώρα έχει το λόγο Κύριε Σμίτα, ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ με την Πρόεδρο και εγώ όταν διάβασα για πρώτη φορά ε, την έκθεση περίμενα κάτι απτό, κάτι συγκεκριμένο ε, και οι πρώτες 26 ε, σελίδες ήταν περιγραφικές όπως είπατε και εσείς. Βέβαια και εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα follow-up και συγκεκριμένα ένας έλεγχος, μια συνοδευτική παρακολούθηση θα έλεγα διότι ε, είναι όλο και πιο δύσκολο να καταλάβουμε την κατάσταση και επιδεινώνεται συνεχώς. Τα είπαν και προλήσαντοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την ε, Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματικά έχουν επιβαρυνθεί πολύ. Αυτό πρέπει να το γνωρίσουμε και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα η κατάσταση επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης ε, και περιμένει κανείς ε, ε, βέβαια με αυτή τη συγχρηματοδότηση και η Ελλάδα και η Ιταλία να ε, συνεργαστούν. Ξέρω ότι δεν υπήρξε συγχρηματοδότηση στην αρχή. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν υπάρχει και καμία παρακολούθηση των επιδόσεων, δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή είναι μια ιστορία μεταξύ εθνικών κρατών της Ένωσης που η μία θέλει να παρέμβει και οι άλλοι δεν μπορούν να δώσουν τα στοιχεία. Πρέπει να έχουμε πραγματικά ανταλλαγή και να μπορούμε να παρακολουθούμε τι μπορεί να βελτιωθεί, τι πρέπει να βελτιωθεί, τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά. Αυτό που ξεχνάμε και πολύ ελαφρά την καρδία μάλιστα πολλές φορές είναι ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους, για ανθρώπινες ψυχές. Η συγγήτρια, κυρία Κινίτση, συμφωνώ και εγώ, είπε ότι υπήρξε αντίδραση, παρκής ανταπόκριση βέβαια σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Πράγματι υπάρχει αυτό το ότι έρχονται για έξι εβδομάδες, ε, αλλά υπάρχουν διαδικασίες πολύπλοκες πριν έρθουν αυτοί και μετά και με τις ε, προσλήψεις και τους διαγωνισμούς. Και ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Αυτό θα βοηθήσει τους πάντες. Γιατί όλοι και οι εκλογείς, ε, οι πολίτες μας βλέπουν ε, πώς αντιμετωπίζει η Ένωση το πρόβλημα. αντιμετωπίζει με επαρκή, με αποτελεσματικό τρόπο. Η έκθεση, η ειδική αυτή, ούτε και για μένα είναι καλή. περιγράφησε Περιγράφει ουσιαστικά τα πράγματα. Τι θέλει η έκθεση, Ποιο είναι ο στόχος, να μας πει ότι ορίστε έτσι τα πράγματα, θέλει να μα εξήσει, αλλά το πρόβλημα, α πούμε, των ασυνόδευτων ανηλίκων. Πώς θα το λύσουμε, το ότι είναι ε, ξεχωριστά τα καταλήματα ε, ή το να είναι ξεχωριστά τα καταλήματα των, για τους ασυνόδευτου ανηλίκου από ότι τους ε, Μα ε, το θέμα είναι οι αρμοδιότητες, είναι κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Σίγουρα είναι καλές και οι συστάσεις, ε, δεν λέω, αλλά θα πρέπει να φροντίσουν να εφαρμοστούν τάχιστα αυτές οι συστάσεις. Πολλές ειδικέ εκθέσεις διατυπώνουν συστάσεις τι κάνουμε, λέμε ναι βεβαίω, τι σημειώνουμε και περιμένουμε μετά χρόνια για να εφαρμοστούν αυτέ οι συστάσει. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά λέω, κατά την άποψή μου, πρέπει να δράσουμε τάχιστα με αυτή την αρχή επικουρικότητα σε εθνικά κράτη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πάψει αυτό το παιχνίδι και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τα hot spot, να υπάρξουν και τα επόμενα βήματα, δηλαδή να βοηθήσουν και τα άλλα κράτη-μέλη ε, και με τη μετεγκατάσταση. Σίγουρα χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά, είναι, υπάρχει ανάγκη διαχείρισης και αν η Ένωση με τους οργανισμούς, με τις ικανότητες και τις αρμοδιότητες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, θα έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κυρία Λαμπάγιοβα, έχει το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι μου λείπουν τα νούμερα, όπως και σε εσά νομίζω και έχω συγκεκριμένα ερωτήματα για κάποιο κόστος. Μου φαίνεται αρκετά περίεργο ότι δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε συγκεκριμένους αριθμούς. Ήδη από πέρυσι, πριν να γίνει η ακρόαση του Επιτρόπου του κ. Βραμόπουλου, είχαμε ερωτήματα και ζητήσαμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος που καταβλήθηκε για τους ε, μετανάστες ανά χώρα. Η απάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και είπε ο Επίτροπος, είναι δύσκολο, παραθέτω, αν όχι αδύνατον, να δώσουμε εκτίμηση κόστους ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των μεταναστών, καθώς η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες, ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον εκπρόσωπο του ε, ελεγκτικού Συνεθρίου, τι γίνεται, τι έχει γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό να μην μπορούμε να δηλώσουμε το κόστος και θα θέλαμε να είναι σαφές αυτό. Και πώς επίσης μπορούμε να το μετρήσουμε σε επίπεδο ανά hot spot. Δεύτερο ερώτημα. Το κόστος της, ε, ε, της πολιτικής επιστροφής. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θέλουν να βοηθήσουν την πολιτική επιστροφής και να κάνουν συγκεκριμένη οικονομική συνεισφορά. Όμως έχουμε τα στοιχεία για αυτό το κόστος αυτής της πολιτικής. Ξέρουμε πόσο καταβάλλεται για αυτή την πολιτική. Σημαντικό. Και τελευταία ερώτηση. Κάτι που, για το οποίο είναι μάλλον ειδικό, ειδική η Κατερίνα Κινέτσι γιατί γνωρίζει για τα παιδιά και τους, ε, ασυνό, τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει διαφορά στο κόστος αν πρόκειται για ενήλικα ε, μετανάστη και για, ε, αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο. Υπάρχει διαφορά. Ενδεχομένως να προσφέρεται αυξημένη βοήθεια ή φροντίδα σε αυτούς τους νέους, τους ανηλίκους. Και δεύτερον, μια δύσκολη ερώτηση για την ηλικία. Γιατί προσωπικά είδα περιπτώσεις στην Ιταλία όπου το θέμα της ηλικίας δεν είναι... Δηλαδή η ηλικία δεν είναι πάντα 18 και αυτό θα άλλαζε το κόστος αν πούμε ότι πρόκειται για όλους όσοι είναι γύρω στα 22 ή μέχρι 22 ετών, θα άλλαζε το κόστος. Λοιπόν, ποιο είναι το κόστος σε αυτήν την περίπτωση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει το λόγο. Επομένω, ξαναδεί, μάλλον δίνω στην κυρία από την γάμα Δέλτα ΧΟΜ. δεν μπορώ να προφέρω το όνομα ακριβώ, ε, μου φάνηκε ελληνικό, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση που υπέβαλε που υποβάλλατε, υποστηρίζουμε την έκθεση της Επιτροπής, τη θέση της Επιτροπής στην παροχή ε, επιπλέον βοήθεια στα κράτη-μέλη και στην Ιταλία και στην Ελλάδα για να βελτιωθεί η κατάσταση στα hot spot και για να γίνει καλύτερη εφαρμογή οποτεδήποτε χρειάζεται. Όσον αφορά τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε όλες τις συστάσεις και η Επιτροπή αλλά και ο οργανισμός θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την πρώτη σύσταση, η Επιτροπή ήδη συντάσσει έναν οδικό χάρτη για να ακολουθήσει αυτή τη σύσταση και για την Ελλάδα και για την Ιταλία. Και στην περίπτωση της Ελλάδας μπορούμε να πούμε επίσης ότι το κοινό σχέδιο δράσης που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών περιλαμβάνει μια διάταξη για να ε, μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις στα νησιά και να ε, επιταχυνθεί η διαδικασία παροχής ασύλου. Όσον αφορά την Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς ενθαρρύνει τις Ιταλικές αρχές να αυξήσουν την δυναμικότητα των hot spot και είναι έτοιμη να υποστηρίξει περαιτέρω τις αρχές. Το, όσον αφορά τους ε, ενηλίκους, υπάρχει μεγάλη ανησυχία εκ μέρους όλων των οργανισμών και της Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βοηθήσει τις εθνικές αρχές για να βοηθήσει να τις βοηθήσει να πλαισιώσουν τους ανηλίκους και στο διορισμό του ειδικού ε, που θα φροντίζει τα παιδιά και να επανδρώσει τα hot spot. Το ίδιο ισχύει και ως τη χρήση ειδικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι οργανισμοί καταβάλουν προσπάθεια να προλάβουν τις ανάγκες που θα εμφανιστούν για τους οργανισμούς, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω τους ειδικού εγκαίρως οποτεδήποτε χρειάζεται. Επιπλέον, οι οργανισμοί εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν ειδικού επιτόπου και για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Όσον αφορά την τέταρτη σύσταση, οι, διαδικασίες, ε, τυποποιημένες ε, διαδικασίες λειτουργίας των ελληνικών ε, hot που ήταν ένα από τα αντικείμενα της σύστασης έχουν προχωρήσει και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Τώρα όσον αφορά την τέταρτη σύσταση για την περιφερειακή δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να της δοθεί θα πρέπει να τεθούν ε, αρμοδιότητες στην Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εντολή έχει ήδη ξεκαθαριστεί στην Ελλάδα στην Ιταλία η κυβέρνηση και οι οργανισμοί και οι Επιτροπή καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να ξεκαθαριστούν να ξεκαθαριστεί ο τρόπος υλοποίησης αυτών των συστάσεων, το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει και τα δύο κράτη-μέλη να ορίσουν έναν υπεύθυνο σε εθνικό επίπεδο για κάθε task force. Όσον αφορά στην πέμπτη σύσταση όπου το δικαστήριο προτείνει να αξιολογηθεί να αξιολογηθούν και να εντοπιστούν ε, τυχόν νομικά και λειτουργικά κενά για να διευκρινιστεί το πώς θα εξελιχθεί το νομικό πλαίσιο αυτής της προσέγγισης των hot spot. Ήδη έχει ξεκινήσει μια πλήρης αξιολόγηση των hot spot και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ελπίζω ότι έτσι σας έδειξα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει, αντιμετωπίζει το δικαστήριο με σοβαρότητα και ότι από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεση έχει αρχίσει να υλοποιεί όλες τις συστάσεις προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει και στο δικαστήριο και στην Επιτροπή σας το ταχύτερο δυνατόν την δράση που θα έχει ολοκληρωθεί. Να έχει... Ενδεχομένως η ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του χρόνου είναι υπερβολικά φιλόδοξη προσδοκία, αλλά οπωσδήποτε το 2018 θα έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις του δικαστηρίου. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα για το πώς, ποια συνέχεια δίνεται και πώς χρησιμοποιούνται τα, χρησιμοποιούνται τα ταμεία. Ακούσατε πέρυσι από τον ε, κύριο Βραμόπουλο, τον Επίτροπο, όταν είχε ε, προσκληθεί στην Επιτροπή, η Κομισιόν δεν είχε λάβει τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Όπως γνωρίζετε, τα ταμεία βρίσκονται υπό κοινή διαχείριση. Λόγω της διαδικασίας της έγκρισης και όλων των ε, των όσων πρέπει να γίνουν με βάση τη ε, νομική βάση στα κράτη-μέλη ε, οδήγησαν σε μια καθυστέρηση στην ε, επίδοση των στοιχείων. Έπρεπε να γίνουν κάποια τεχνικά βήματα ώστε να μπορεί η ελεγκτική αρχή να, να οριστεί η ελεγκτική αρχή των ταμείων αυτών. Όταν λοιπόν ε, ήρθε στην Επιτροπή σας ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος, είχε λάβει λίγα μόνα στοιχεία επί των οποίων θα με τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση. Το Μάρτιο του 2017 λάβαμε τα στοιχεία του 2016 και η απόφαση για την εκαθάριση των λογαριασμών του 2016 θα ληφθεί αφού αναλυθούν τα στοιχεία και, τα, ε, ε, με βάση αυτά που θα μας δώσουν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, σχετικά με το πραγματικό κόστος ε, των, με, των μεταναστών, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να απαντήσω. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει ε, να κάνει την ανάλυση στο εσωτερικό του κράτους μέλους για το πραγματικό κόστος κάθε μετανάστη. Θα μελετήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε το ταχύτερο δυνατόν. Το κόστος της, της πολιτικής επιστροφής, μάλλον για το κόστος αυτό, δυστυχώς ισχύει το ίδιο. Δεν Δεν ε, γνωρίζουμε αν είναι δυνατό να το υπολογίσουμε αυτό με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορά κόστους, ε, αν, ε, ανάλογα αν πρόκειται για μετανάστη ή ανήλικο, είναι σαφές ότι υπάρχει διαφορά, διότι περισσότεροι πόροι δαπανώνται για τους μετανάστες για, που είναι ανήλικοι και από το κράτος μέλος και από τους οργανισμούς για τη φροντίδα των ε, ανηλίκων. Άρα ο προπολογισμό ε, θα είναι υψηλότερος γιατί παρέχονται περισσότερες ε, υπηρεσίες. Κατά τα άλλα δεν γνωρίζω αν η Κομισιόν είναι σε θέση τη στιγμή αυτή να κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στο κόστος ε, του ενηλίκου και του ανηλίκου. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Αν όχι, παρακαλώ ζητήστε μου να επανέλθω. Μάλιστα σε ό,τι αφορά το τυπολιπόταν των προσδοκιών μα ε, η ειδική έκθεση εξακολουθεί να υπολείπεται. Για τον Επίτροπο Αβραμόπουλο που ήταν για τη διαδικασία απαλλαγή, ε, μάλλον που θα τον δούμε για τη διαδικασία απαλλαγή, θα το συζητήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη σύσταση για του ασυνόδευτού ανηλικου συγκεκριμένα. Υπάρχουν επιτρόποι ανηλίκων σε ε, όλα τα hot spot, ναι ή όχι. Δεν το κατάλαβα ε, μπορείτε να μου το διευκρινίσετε. Υπάρχει έστω ένας ε, υπεύθυνο ε, για το να σε κάθε κέντρο ταυτοποίησης. Ε, the, the appointment... Σε σχέση με την Ιταλία, ο διορισμός του αξιωματικού προστασίας του παιδιού για έναν ασυνόδευτο ανήλικο ε, σχεδόν ε, ολοκληρωθεί από τις Ιταλικές αρχές. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που σχετίζεται με αυτή την προσπάθεια κατόπιν ε, της έκθεσης της οποίας η Δεξικομισιόν για να διαθεωρηθεί η κατάσταση στην Ιταλία και για την Ελλάδα τώρα. Έχει διοριστεί ε, ο αρμόδιος προστασίας του παιδιού από τις ελληνικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείται σχεδόν. Ε, it means that... σημαίνει ότι αναμένουμε οι τελικές αρχές να διορίσουν τον αξιωματούχο προστασίας το παιδιού τον επόμενο μήνα. Also dann nächsten Monat, ich gehe davon aus, dass es nicht das spanische Manana ist. Μάλιστα. Όταν λέμε τον επόμενο μήνα, όντως μιλάμε για τον επόμενο μήνα, όχι για ένα ισπανικό αύριο. Αναφέρατε ότι θα μας ε, δώσετε και μία έκθεση και ότι θα μας πείτε και ποια είναι η προθεσμία για την παράδοση της έκθεσης αυτής. Φυσικά όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ε, γιατί είμαστε πολιτικοί. Ναι, ναι, ναι, θα το εξηγήσω αυτό αργότερα. Παρακαλώ, κύριος Βέσπα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να απαντήσω σε ακούστηκαν στη συζήτηση. Να ξεκινήσω με το αντικείμενο του ελέγχου και εμείς στο λεκτικό συνεδρίο κατά τη ε, διάρκεια των εξητών ε, που είμαι εδώ κάναμε κριτική στον εαυτό μας ότι καθυστερούσαμε στην παράδοση των εκθέσεών μας. Και αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε υποβάλει μία έκθεση, όταν υποβάλουμε μία έκθεση για έναν έλεγχο, ήδη το θέμα δεν είναι πλέον πολιτικά καυτό. Αυτή την εντύπωση έχω τέλος πάντων ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασκήσει τέτοια κριτική σε εμά. Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε αυτό, λειτουργώντας κάπως ταχύτερα και κάνοντας πιο συγκεκριμένους ελέγχους, έτσι ώστε να είμαστε πιο γρήγοροι. Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στο στα θέματα που είναι σημαντικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε τον έλεγχο αυτό, ε, μιλούσαμε για ανθρωπιστική καταστροφή, για, όταν μιλάμε για το πώς χειρίστηκαν ε, το προσφυγικό τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε το 2015 στην προσέγγιση των ε, hot spots, των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Αυτό ήταν το πιο καυτό θέμα τότε. Τώρα, πρέπει να δείτε το θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού ως μια ολόκληρη αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή ξεκινά με την πραγματική διαχείριση της ροής των μεταναστών, διευκολύνοντας την πλήρη ταυτοποίηση, καταγραφή και δεκτυλοσκόπηση των μεταναστών. Χωρίς αυτό τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Καμία χώρα δεν ε, θα δεκτεί τη μεταγκατάσταση των μεταναστών χωρίς να έχει υπάρξει πριν αυτή η διαδικασία στην αλυσίδα. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε εκεί και οι απαντήσεις μας ήταν σαφείς. Τα hot spot ε, πράγματι βοήθησαν ε, να επιληθούν καταστάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ξεφύγει και επίσης αποτελούσαν τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα, την καταγραφή δηλαδή. Το μεγάλο μας πρόβλημα βεβαίως ήταν ότι καθώς ήταν ταχύς ο έλεγχος αυτός, μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι δεν θα είχαμε πλήρως στη διάθεσή μας όλες τις απαραίτητες οικονομικές πληροφορίες. Ε, η Κομισιόν μας έδωσε τα στοιχεία το Μάρτιο φέτος, όμως είχαμε ήδη ολοκληρώσει εμείς τον έλεγχό μας. Δεν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, ήταν αδύνατο να κάνουμε οικονομικό έλεγχο. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια σε έναν επόμενο έλεγχο ή θα μπορούσαμε να κάνουμε ελέγχους που αφορούν το υπόλοιπο τμήμα της αλυσίδας. Να τονίσω ότι όταν ε, υλοποιήσαμε αυτόν τον έλεγχο, δεν ε, είχαμε οικονομικές πληροφορίες για την Ελλάδα η Ιταλία δεν είχε καν ζητήσει κονδύλια τότε. Και νομίζω ότι αυτό είναι σχετικό όταν το συζητούμε αυτό. Γιατί επιλέξαμε στενό αντικείμενο λόγω της σημασίας του και για να μπορούμε να δημοσιεύσουμε συστάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σχετικά γρήγορα στη συνεχιζόμενη διαδικασία της hot spot Και εγώ νομίζω ότι ήταν καλή η απόφαση αυτή. Και όπω μας έδειξαν οι πρόσφατε εξελίξεις, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περισσότερα hot spot Αυτό το δείξαμε στην έκθεσή μας. Κάτι που σίγουρα προσέξαμε ήταν το εξή. Όταν υλοποιήσαμε αυτόν τον έλεγχο δεν ε, υπήρχαν ε, επίτροποι προστασίας του παιδιού. Τώρα έχουμε την ενημέρωση από την Κομισιόν ότι επιλύεται αυτό το πρόβλημα. Όμως αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που θέλαμε να συστήσουμε και νομίζω ότι η δική μας έκθεση βοήθησε την Κομισιόν στο συνεχιζόμενο έργο της για να βελτιώσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι ε, υπάρχει αυτή η, το δίλημα, θέλετε και αυτή η διαφορά, ε, μια ειδική έκθεση που ουσιαστικά έχει καθαρά ιστορικό χαρακτήρα και μια ειδική έκθεση η οποία ε, εξελίσσεται και τα στοιχεία μεταβάλλονται. Μπορείτε να μας δώσετε όμως κάποια προθεσμία. Ναι, Όλες οι ειδικέ εκθέσεις έχουν το follow-up. Υπάρχουν δηλαδή πάντοτε εκθέσεις ε, μέσα σε τριετία νομίζω εκεί η Ροπολή γίνεται αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ ως μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου που θα σας πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη όχι για follow-up αλλά και έλεγχο, audit κανονικό γιατί αλλάζουν τα πράγματα όπως είπατε και θα πρέπει να ελέγξουμε τα, τα στοιχεία όπως πάνω χάρη το κομμάτι που αφορά την κατάσταση. Άρα θα ξεκινήσει μάλλον ένας νέος έλεγχος. Τώρα πότε δεν το ξέρω. Η δική μου εντολή λίγη 1η Μαρτίου. Ε, η θητεία μου λίγη και δεν ξέρω αν θα έχω εκ νέου την αρμοδιότητα Σίγουρα για του χρόνου όμως το ελληνικό συνέδριο κατά προτεραιότητα θα ασχοληθεί με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κινίτσι, ποιος από τους δύο εισηγητές για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, κύριε Κινίτσι, πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες τις συνεισφορές στη συζήτηση. Γιατί η αναμφισβήτητα μας έδειξαν ε, ουσιαστικά ποιο είναι το αντικείμενο του ελέγχου. Και χαίρομαι που πρόσωπο του λεκτικού Συνεδρίου μας μίλησε για τη δυνατότητα ενός νέου ελέγχου που θα διερευνήσει προσεκτικότερα το χρηματοοικονομικό ζήτημα, γιατί σίγουρα χρειάζεται και εμβάθυνση για το κόστος. Όπως επιβεβαιώθηκε και από την εκπρόσωπο της Κομισιόν σε ό,τι αφορά ιδίως την Ιταλία. Πράγματι, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για να ακολουθήσουμε το περιεχόμενο των συστάσεων. Και γίνεται και ιδιαίτερη προσπάθεια στο θέμα των ασυνόδευτων ενηλίκων. Ακριβώς ε, προβλέπουμε το διορισμό εμπειρογνωμόνων, ειδικών για την υποδοχή των ευάλωτων ανηλίκων. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ερωτήσεις της κυρίας Δαμπάλοβα όπως ε, αναφέρθηκε στο θέμα των ανηλίκων ε, και φυσικά στο οποίο εγώ είμαι ειδικός όπως ε, υπόθηκε. Το θέμα του κόστους θα το δούμε στο μέλλον. Όμως οι ενήλικοι χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία και μεγαλύτερη υποστήριξη και περισσότερες υπηρεσίες. Δηλαδή χρειάζεται νομική προστασία, σκεφτόμαστε στο διορισμό επιτρόπων, αλλά και προστασία ψυχολογικού τύπου, ψυχολογική υποστήριξη, προστασία της υγείας τους και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια πιο πλήρης προστασία από ότι στην περίπτωση των ενηλίκων. Τώρα για το πρόβλημα των ε, της ηλικία. Ε, κοιτάξτε, κάποιος θεωρείται ανήλικος ε, κάτω από το 18. Στη χώρα μου προβλέπεται η προστασία μέχρι το 18, όμως κατόπιν γίνεται μία προσπάθεια να μην διακοπεί αυτή η υποστήριξη, αυτή η προστασία όταν κάποιος κλείσει τα 18. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο. Στους ποινικούς, στα ποινικά ε, όργανα, ε, παραδείγματο χάρη, θεωρείται κάποιος ανήλικος μέχρι τα 25 για να μην διακοπεί ή μια εκπαιδευτική διαδικασία που μπορεί να έχει ξεκινήσει. Αυτό γίνεται στη χώρα μου γενικά για την προστασία των ανηλίκων. Γιατί ξαφνικά να εγκαταλείψουμε έναν ανήλικο ο οποίος ε, είχε προστασία, είχε πίτροπο και είχε όλη την υποστήριξη να εγκαταλειφθεί όταν ε, κλείσει τα 18 και ξαφνικά να μην έχει καμία προστασία και υποστήριξη σημαίνει ότι θα τον εκτέσουμε σε μια κατάσταση κινδύνου γιατί κλείνει τα 18 και απλά γίνεται αυτό σε μία μέρα. Δηλαδή αν κάποιο είναι 18 και μία μέρα δεν έχει καμία διαφορά από την προηγούμενη μέρα. Έτσι, λοιπόν, ε, το χάρη αν, ε, ε, αν κάποιος είναι ανήλικος, προσπαθούμε να βρούμε μια οικογένεια για να υποδεχτεί τον ανήλικο. Η προσπάθεια λοιπόν ε, για να μην διακοπεί η προστασία γίνεται ακόμη και αν ε, ενηλικιωθεί το παιδί. Έτσι, λοιπόν, σίγουρα σε σχέση με το κόστος ε, θα είναι σκόπιμο να γίνει μια περαιτέρω έρευνα, γιατί όλοι καλούμαστε να καταβάλουμε οικονομική προσπάθεια, όχι μόνο η Ιταλία, αλλά και άλλες χώρες και κάτι τελευταίο. Είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή έχει φωτογραφίσει μια συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό αφορά τη στιγμή μιας διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει και άλλα βήματα όπως είναι παραδείγματος χάρη, μεταγκατάσταση κτλ. Πάντως ε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι μας βρίσκει καλούς σύμφωνους. Ο κύριος De Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι όταν καταρτήσαμε το έγγραφο εργασία, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη του περιορισμού του ελεγκτικού συνεδρίου, όπω ακούσαμε και εδώ. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι το βλέπετε και με τις δικές μας συστάσεις, τις έχουμε λάβει υπόψη αυτές τις, ε, αυτά τα προβλήματα στους περιορισμούς, γι' αυτό και ζητούμε follow-up συμφωνώ ότι για ένα χρηματοοικονομικό έλεγχο ε, χρειάζεται αυτό να μπει ως τόπο προτεραιότητα. το είπε και ο κύριος Βέσπεκ. Το κόστος επίσης είναι σημαντικό. Και τα νούμερα λείπανε. Γι' αυτό και αυτή η ειδική έκθεση διαφοροποιείται από άλλες ειδικές εκθέσεις. Δηλαδή δεν ήταν δυνατό κατά πόσα πιθανότητα από ό,τι φαίνεται να γίνει αυτός ο χρηματοοικονομικός έλεγχος στην προκειμένη περίπτωση και προς την Κομισιόν. Ε, στρεφόμενος να πω ότι η Επιτροπή μας ε, έχει ε, πολλές πολύ σημαντική δουλειά μπροστά τη και σε ό,τι αφορά την απαλλαγή τη Κομισιόν. Μιλήσατε για τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και για τη συνάντηση που θα έχουμε. Μετά από τη συζήτηση αυτή όμως σήμερα διαρωτώ με μήπως και ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς θα έπρεπε να συμμετέχει που δραστηριοποιείται ενεργά και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και επειδή τα πράγματα έχουν σοβαρέψει στην προηγούμενη περίπτωση και την μας Επιτροπή και ενεργοποιείται όταν σοβαρεύουν τα πράγματα ο κ. Τίμερμαν, θα πρέπει να τον καλέσουμε. Η Κομισιόν έχει μόνο μερικές πληροφορίες, ε, τμηματικές δηλαδή. Ε, μας λείπει η εικόνα, η ολόκληρη εικόνα και δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εξαψήφιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρατήρηση ε, για το κόστος του μετανάστη. Τι να σας πω, αμφιβάλλω ότι κάτι τέτοιο είναι λογικό. Ε, γιατί πράγματι είναι πολύ παραγοντικός υπολογισμός, η ένταξη, η εγκληματικότητα, μεγάλο φάσμα, πλήρες φάσμα. Αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι βέβαια το κόστος του κάθε κρίκου της αλυσίδας. Δηλαδή υποδοχή στην εγκατάσταση, εξέταση της αίτησης, ε, επιστροφής. Το κόστος κάθε σταδίο αυτού. Αυτό μάλλον εννοούν οι συνάδελφοι που μίλησαν για το κόστος μετανάστε, Πιο στοχευμένα. Και τελευταία παρατήρηση. Υπάρχει διαφορά. Το κόστος επιστροφής μπορεί να είναι τεράστιο. Να μην ξεχνάμε όμως πως όταν βλέπεις όλη την αλυσίδα η επιστροφή είναι το ίδιο σημαντική με την ε, εισδοχή των ε, προσφύγων και η δημόσια υποστήριξη. την υποδοχή μεγάλων αριθμών προσφύγων και μεταναστών εξαρτάται και από το πόσο αποτελεσματικές είναι οι επιστροφών. Το ένα πάντα σχετίζεται με το άλλο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να φτάνουν συνεχώς ε, οι λαδομετανάστες στην Ιταλία ε, δεν είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές γι' αυτό. Το θέμα δεν είναι τόσο το κόστος, όσο η αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ερχόμαστε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης που είναι μια γνωμοδότηση θα μας την παρουσιάσει ο συνάδελφος Φλάναγκαν για το BBI, Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων. Ο συνάδελφος Φλάναγκαν, παρακαλώ, παρουσιάστε μας την ομοδότησή σας. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κοινή επιχείρηση βιομηχανικών βιοπροϊόντων δημιουργήθηκε το 2014 για 10 χρόνια με την πρωτοβουλία της κοινοπραξίας βιομηχανικών βιοπροϊόντων συμμετέχουν αφενός μεν η, Ένωση που εκπροσωπείται από την Επιτροπή και αφετέρου η ε, Κοινοπραξία Βιομηχανικών Βιοπροϊόντων. Είχε συμφωνηθεί ότι η ε, BIC θα, ε, ε, θα είχε συνεισφορά τριεπλάσια από τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εταιρείε όμως ε, που συμμετέχουν στην BIC κατανοητά είναι, διστάζουν να συμμετέχουν ε, στη χρηματοδότηση του προβλήματος γιατί κατά κάποιο τρόπο αισθάνονται ότι χρηματοδοτούν τους ανταγωνιστές τους. Όμως ε, θα ήθελα να μπορούν να ε, χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες, οι οποίες ενδιαφέρουν. Υπό την ε, παρούσα νομική βάση αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι όμως πάρα πολύ απλό να ληφθεί απόφυση για να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή και να υποστηριχθεί από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόρχλ έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάνακαν εξήγησε τους, ε, τον χρηματοοικονομικό μηχανισμό που λειτουργεί στην BBI. Ε, Ήμουν εισηγητής. Άκουσα πολλέ ε, παρατηρήσεις από διάφορες πλευρές και νομίζω ότι αυτή είναι η καλή λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Αν περάσει από την Ολομέλεια και εγκριθούν από το Συμβούλιο αυτές οι αλλαγές, η, η χρηματοοικονομική συνεισφορά, η χρηματοδοτική συνεισφορά θα αλλάξει. Ο ιδιωτικό τομέας θα μπορεί να πληρώνει, να, να καταβάλει χρήματα σε επίπεδο προγράμματος. Μέχρι στιγμής ε, έχει καταβληθεί μόνο ένα εκατομμύριο από τα 182 εγώ έχοντας μελετήσει όλες τις εναλλακτικέ είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Πρέπει να κινηθούμε προσεκτικά για να δούμε πώς ε, δρούν αυτές οι επιχειρήσεις και να τα λάβουμε υπόψη μας κατά την απαλλαγή. Η αλλαγή στους κανόνες χρηματοδότησης σε επίπεδο έργου θα εξαρτηθούν επίσης από το αν οι εταιρείε θα εκπληρώσουν Πλήρω τις υποχρεώσεις τους. Και η Επιτροπή μας θα είναι η πρώτη που θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όντως έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές και ότι έχει γίνει αλλαγή στη συμπεριφορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φλάναγκαν όσον αφορά τη γενική προσέγγιση στο θέμα. Είναι σωστό. Και θα πρέπει η νέα μορφή χρηματοδότησης που τώρα προτείνει η Κομισιόν να υποστηριχθεί από εμά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται το δυναμικό των επιχειρήσεων να συνεισφέρουν. Στο παρελθόν ήταν στα πλαίσια ενός γενικού πλαισίου που δεν ικανοποιούσε όλες τις επιχειρήσεις γιατί δεν έβλεπαν ποιο ήταν το πλεονέκτημα στο να προχωρήσουν. Πέραν αυτού υπάρχουν και κάποια ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να φανούν στην έκθεση. Πρώτον, γιατί διάβασα την πλήρη απόφαση της Επιτροπής και την ε, λογική που τη διέπει η κίνηση που προέρχεται από πλευράς Επιτροπής είναι το, το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας, όπως λένε. Διαβουλεύτηκαν με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιστεύω ότι έχουν, μπορούμε πολλά να μάθουμε από αυτό. Αν ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που δύναται να αποδώσει, είναι απολύτως απαραίτητο η Κομισιόν να συνεργαστεί. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε όχι μόνο στο πλαίσιο της, ε, των βιομηχανικών βιοπροϊόντων, αλλά και σε όλους τους τομείς. Δεύτερον, εάν αυτό είναι αποτελεσματικό και αν απελευθερωθεί το δυναμικό που έχουν επιχειρήσεις για να συνεισφέρουν περισσότερο, το θέμα είναι τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό για άλλες κοινέ επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να γνωρίζουμε. Από τη μία πλευρά μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή, όπως ακούσαμε, από την άλλη μπορεί να απελευθερωθεί δυναμικό και σε άλλους τομείς. Θα ήθελα αυτό να αναφερθεί στην έκθεση και θα φροντίσω να το ε, συμπεριλάβω. Από την άλλη πλευρά, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα επανέλθει το θέμα σε εμά. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο από πλευρά των κοινών επιχειρήσεων να σκέφτονται τι έχουν μάθει συνεπή αυτής της αλλαγής στις ετήσιες αναφορές τους. Εμείς θα το ξαναεξετάσουμε αυτό του χρόνου νομίζω και τώρα θα πρέπει να επισημάνουμε στις παρατηρήσεις μας για την έκθεση αυτή ότι είναι ανάγκη οι κοινέ επιχειρήσεις από μόνες τους να σημειώνουν ποια είναι για αυτούς τα επιχειρήματα ποια είναι η αξία που προσφέρουν στους πολίτες και στους φορολογουμένους. Θα πρέπει αυτά τα θέματα από τώρα να περιληφθούν και να τεκμηριωθούν όταν θα γίνει η πλήρης αξιολόγηση των κοινών επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα τέσσερα θέματα που θα ήθελα να εμφανιστούν στην έκθεση και θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες σε συνεργασία με τον κύριο Φλάνγκαν. Το βασικό θέμα για την Επιτροπή μας είναι αν προχωρήσουμε στο δρόμο αυτής της αλλαγής που το δέχομαι είναι απαραίτητη, είναι προφανής όπως είπε και ο εισηγητής, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα ωφέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντλαμπάγιοβα. Συμφωνώ με το εισηγητή και τους και εισηγητές ότι ε, η προθεσμία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, τα μέλη του BIC να την τηρήσουν. Ε, συμφωνώ λοιπόν και καλό είναι να υπάρξει μια γενική επισκόπηση Είναι πολύ καλή η ε, γνωμοδότηση και συμφωνώ επίσης ότι με τις τροποποίησεις της Κομισιόν θα υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για χρηματοοικονομικές συνεισφορές και από άλλες πηγές και όχι μόνο από τον προϋπολισμό της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Αλαφράγκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή την ανάλυση συγητή όμως ε, η πραγματικότητα είναι βάση των αποτελεσμάτων της επιχειρήσης που δημιουργήθηκε βάσει ενός κανονισμού του 2014 μας δείχνει ότι δεν έχει λειτουργήσει. Δηλαδή, αν ε, δει κανείς την πρόβλημα ο ήταν ε, ότι η κοινοπραξία θα συνεισέσφερε 182,5 εκατομμύρια, ενώ έχει συνεισφέρει 0,5 μόνο. Η Κομισιόν έχει αναστείλει τη δική της συμμετοχή, καθώς ε, η κοινοπραξία δεν ε, συνεισέφερε. Η Κομισιόν έπρεπε να συνεισφέρει 70 εκατομμύρια και έχει αναστείλει τη δική της ε, συνεισφορά. Νομίζω λοιπόν είναι σημαντικό, Πρόεδρε, να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε η κοινή επιχείρηση και γιατί ο κανονισμός δεν έχει παράξει τα αποτελέσματα που είχε θέσει. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι τελικά θα δώσουμε την εξής εντύπωση ότι ουσιαστικά θα συγχωρήσουμε αυτή την ε, συνεισφορά 182,5 εκατομμύρια και τελικά αν ε, θέσουμε την ε, συνεισφορά του αναέργο ε, τελικά τι θα κάνει η κοινοπραξία απλά θα συνεισφέρει εκεί όπου θεωρεί ότι μπορεί να έχει κέρδος. Εγώ δεν είμαι αντίθετο ακριβώς στην πρόταση του συγητή, αλλά θα ήθελα ξεκάθαρα να δω γιατί αυτό δεν έχει λειτουργήσει και αν όλα είναι τόσο απλά όπως απλώς να γίνει ε, μια τέτοια τροποποίηση του κανονισμού, αρκεί αυτό για να λειτουργήσει. Και θα ήθελα να μου πείτε ποιε είναι οι συνέπειες της έλλειψης αποτελεσματικότητας ε, τη επίτευξη των στόχων του κανονισμού που δημιουργεί την ε, κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων. Ουσιαστικά αυτό που θέλω εγώ είναι τελικά τι θα κάνουμε. Απλώ θα διευκολύνουμε την άδειξη μεγάλων επιχειρησιών σε ένα σχέδιο à la carte εδώ βλέπουμε με σαφήνεια ότι δεν έχει λειτουργήσει αυτό το σχέδιο και αναρωτιέμαι αν αρκεί να κάνουμε μια τροποποίηση του κανονισμού έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό το consortium να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές. Αλλά ήθελα να ξέρω αν αυτή η νέα τροποποίηση του κανονισμού, αυτή η νέα διαδικασία σημαίνει ότι θα συνεχίζει να έχει την υποχρέωση το κονσόρσιουμ να συνεισφέρει αυτά τα 182,5 εκατομμύρια. Ξέρετε, σε μισή ώρα έχουμε την κοινή συνεδρίαση προπεριβάλλοντος, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι. Ζήτησε ο κύριος Χέης τον λόγο. Ναι, πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Διάβαζα την ε, έκθεση της Κομισιόν την αρχική και από ό,τι κατάλαβα τότε δεν υπάρχει μελητή αντικτύπου. Θα πρέπει να μας εξηγήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδομένου του ποσού, ε, του ύψους του ποσού για τον οποίο μίλησε και ο προλογηγούμενος ε, ε, ε, πρέπει να μας εξηγήσει ξεκάθαρα η Κομισιόν. Κυρία από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνα. Αν μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλή σας ημέρα. Η πρωτοβουλία BPI φτάνει σχεδόν στο μέσο του κύκλου Η μόχλευση αυτό το 16 υπολογίστηκε ήδη σε 2,6 δηλαδή ένα ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης αντιστοιχεί σε 2,6 ιδιωτικής χρηματοδότησης ήδη. Και αυτό είναι πολύ κοντά στο αναμενόμενο επίπεδο αποτέλεσμα μόχλευσης που το έχουν υπολογίσει 2,8 για το τέλος αυτής της ε, περίοδου. Και είναι από τις 7 κοινοπραξίες ε, που λειτουργούν στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 το υψηλότερο. Άρα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ιδιωτικής βιομηχανίας. σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές ε, εισφορές. Ε, σίγουρα αυτό αυξάνει το επίπεδο της μόχλευσης, ε, αυξάνει τις επενδύσεις για απασχόληση, για μια κοινωνία μετά το πετρέλαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα έχει αναστείλει, όχι περικόψει, έχει αναστείλει με εκατομμύρια τη συνεισφορά για την ε, προάσπιση των χρηματοοικονομικών συμφέροντων περιμένοντα την τροποποίηση και θέλω να σα ευχαριστήσω τον κύριο Φλάναγκαν συγκεκριμένα για την θετική αυτή νομοδότηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπει και προσέχει πολύ την παροχή των ε, χρηματοδοτικών εισφορών της βιομηχανίας. Και με, χάρη, με την τροπολογία αυτή, ελπίζω, θα έχουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο συντελεστή μόχλευσης από ό,τι τώρα. Σε ό,τι αφορά την κλίμακα της βιομηχανίας. 120 εκατομμύρια είναι το ποσό για τις ΜΜΕ. 30% της συνεισφοράς της Ένωσης. Υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο του ορίζοντα 2020. Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στα ερωτήματα και να καρδιασκέσα τις ανησυχίες. Πρόεδρος. Δυστυχώς όμως ε, πρέπει να συνεχίσουμε και επειδή έχουμε και άλλα θέματα, δώσω τον λόγο στον κύριο Φλάνδη για να κλείσει. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Ε, ξέρετε, ε, όπως κοιτάς το κενό πριν επιδείξεις, ε, τώρα και αυτό κάνουμε. Ε, κοιτάμε το άλμα που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας. σίγουρα ε, νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε συμφωνήσει ε, δημοσίως. Ε, βέβαια, ξέρω ότι κάνετε τη δουλειά σας, συνάδελφε. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Μέχρι αύριο στις 12 είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Έτσι λοιπόν, υπομονώ να τις λάβω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. 4 Σεπτεμβρίου θα ασχοληθούμε εκ νέου με την ψηφοφορία και ελέγξτε το με την γραμματεία ε, αν θέλουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, διότι είναι πολύ πιεστικό το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πηγαίνω στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για μία έκθεση follow-up που έχετε μετά την ειδική έκθεση παριθμών 9 του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την έψο δηλαδή την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων επιλογής προσωπικού. Θέλω να σας δώσω, κύριε Διευθυντά της ΕΨΟ, κύριε Μπέρφιλ, τη δυνατότητα να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα, αν έχουν βελτιωθεί. Ε, ξέρω ότι επιβαρυνθήκατε στην αρχή με ένα κακό, με μια κακή έκθεση, με μια κακή διακή έκθεση. Για να μας πείτε τώρα αν τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το τι κάναμε και κάναμε πολλά ε, τα τελευταία δέκα χρόνια, πρέπει να σας πω, εστιάζοντας τις πολύ χρήσιμες ε, συστάσεις ε, της ειδική έκθεση του Εκτικού Συνεδρίου για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της ΕΠΣΟ. Sorry, What we have done is... Αυτό που έχουμε κάνει λοιπόν στην ε, ΕΠΣΟ είναι ένας ριζικός μετασχηματισμός των εργασιών μας και εστιάσαμε σε τέσσερις τομείς που ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις ε, ε, συστάσεις του Συμβουλίου. Πώς σχεδιάζουμε τις ανάγκες, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, τις ε, δοκιμασίες, των τον επαγγελματισμό και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ταλαντούχους ε, υποψηφίους ε, και να προωθήσουμε και τη διαφορετικότητα. Η πρώτη σύσταση έλεγε ότι δεν είχαν ε, επικοινωνήσει, δεν είχαν δώσει έγκαιρα οι θεσμοί τις ανάγκες τους για στελέχωση. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι ότι έχουμε το στρατηγικό πλέον σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους. Δεν είναι τέλειο το σύστημα, αλλά μας βοήθησε να καταλάβουμε περισσότερο τα, τη σχέση προσφοράς ζήτησης. Και επίσης έχουμε και κάποιους ετήσιους κύκλους ε, ε, διαγωνισμών, γιατί επανέρχονται οι ανάγκες ε, και καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο πιο ορθολογικά τους πόρους μας και αυτοί οι θεσμοί που ουσιαστικά έχουν σε τακτά διαστήματα ανάγκες να μπορούν να τις καλύπτουν. Ε, τριετής είναι ο κύκλος στρατηγικού σχεδιασμού, κάθε χρόνο προσαρμόζεται και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Το βλέπετε και στην επόμενη διαφάνεια, ε, στην πράξη πώς λειτουργεί το σύστημα. Τρεις βασικοί κύκλοι διαγωνισμών ετησίως υπάρχουν. Είναι σταθερά τα χρονοδιάγραμματα από το 2010 και μετά. Οπότε είμαστε και πιο παρόντες στην αγορά προσλήψεων, γιατί ξέρουν πού να αποταθούν οι δυνητικοί υποψήφοι. Έχουμε λοιπόν διοικητικού υπαλλήλου στην Άνοιξη, γλωσσομαθεί το καλοκαίρι και στα τέλη του χρόνου βοηθεί συνεργάτες. Και στα κενά που μένουν έχουμε εξειδικευμένους διαγωνισμούς. Δεύτερη σύσταση που έλεγε ότι είναι πολύ μακρά χρόνια διαδικασία επιλογή προσωπικού. Ναι, είναι ακόμη και μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο διάρκεια. Υπάρχουν όμω και υποχρεώσει για του ε, εργοδότε δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, πρέπει να του αντιμετωπίζουμε όλου με δίκαιο τρόπο, ισότιμα και να λάβουμε σωστέ αποφάσει, εφόσον πολλέ φορέ προσφέρουμε διαβίου απασχόληση. Έχουμε μειώσει όμω το χρόνο ε, του ε, προσωπικού κατά 6% και πολλέ φορέ και περισσότερο. Εδώ βλέπετε ένα πάρα πολύ αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα ε, πριν από το 2009-2010, οπότε και εφαρμόστηκε η νέα διαδικασία. Βλέπετε τότε ότι ένας διαγωνισμός θα διακουσε δύο χρόνια και οι επιτυχόντες ε, είχαν 50 δυνατότητες να προσληφθούν ή και χρόνια ολόκληρα. Τι κάναμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα αλλάξαμε τη διαδικασία επιλογής. Από δύο χρόνια πλέον είμαστε στους 9 ε, με 12 μήνες και με τα θεσμικά όργανα προσπαθήσαμε να καταστήσουμε την όλη διαδικασία πιο διαφανή και ταχύτερη. Φέτος τώρα, 5 Ιανουαρίου, κάναμε μια ριζική αλλαγή στις διαδικασίες ε, πρόσληψης. Μεγάλο ε, μέρος του προσωπικού ε, μπορεί να προσβληθεί πολύ γρήγορα, ιδίω στην Κομισιόν. Και το σύστημα αυτό είναι πολύ πιο οικονομικό, πολύ πιο ταχύ σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Το 2000 ήταν τελευταία δικασία, είχαμε 30.000 για γενικό διαγωνισμό, 10.000 πέρασαν και μόνο κάποιες εκατοντάδες προσλήφθηκαν. Δεν είναι και το βάλει φορμάνι και πολύ καλό. Έχουμε ένα πολύ καλύτερο τώρα σύστημα. Δηλαδή έχουμε μια μόνιμη πρόσκληση υποβολή ε, εκδήλωση ενδιαφέροντο. Και δεν του ελέγχουμε όλου. Έχουμε ένα εργαλείο όπου hiring manager μπορεί να εξετάσει όλες τις αιτήσει ε, και να βάλει σε έναν κλειστό κατάλογο, σαν κατάλογο προεπιλογής, ε, αυτούς του οποίου θέλει μετά να τους κάνει συνέντευξη. Και μόνο αυτοί οι οποίοι θα περάσουν από συνέντευξη θα προσληφθούν ελέγχονται. Όποιοι περάσουν αυτό το τεστ δεν χρειάζεται να το ξαναπεράσουν, γιατί παραμένει το σκορ που πέτυχαν για 10 χρόνια. Και μπορεί να ξαναδοκιμάσει αν αποτύχει μετά από 6 μήνες. Άρα έχουμε μια δεξαμενή ατόμων που ήδη έχουν δοκιμαστεί και δεν χρειάζεται λοιπόν ένας-δύο χρόνια για τα ε, για τους 30.000, μπορούμε να τους επιλέγουμε τους συμβασιούχους μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Η επόμενη σύσταση, η κριτική του ηλεκτρικού είναι ότι δεν επιλέγουμε όλους αυτούς που έπρεπε να επιλέξουμε. Και πολύ σωστά ε, τα είπαν στο ηλεκτρικό στρατό Το 60% μόνο είχαμε επιλέξει μετά από μια διαδικασία δύο ετών σε ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό. Εδώ βλέπετε πώς με το στρατηγικό σχεδιασμό και τις καλύτερες διαδικασίες επιλήξης πώς έχει αλλάξει δραματικά η κατάσταση. 2016, 99,7% ε, ήταν ο στόχος, ε, που ο στόχος ήταν το 120% και εμείς πετύχαμε το 99,7% άρα μπόρεσαν να διαλέξουν όλους όσους χρειάζονταν. Επίσης καταφέραμε να πείσουμε τα θεσμικά όργανα το σύστημα του flagging να το ε, καταργήσουν, όπου ουσιαστικά τους μπλοκάριζαν ε, τους υποψηφίους για ένα χρόνο. Αυτό πάει τώρα. Έχουμε ε, ελεύθερη αγορά. Και επειδή οι θέσει που χειρεύουν δημοσιεύονται, ηλεκτρονικά, υπάρχει ισότιμο πίεδο ανταγωνισμού και οι υποψήφοι επιτυχώντε ε, όπου και αν είναι μπορούν να υποβάλλουν για αυτές τις ε, θέσεις που είναι ανοιχτέ με διαφανή τρόπο. Γεωγραφική εξορρόπηση επίσης είναι ένα δύσκολο θέμα και σίγουρα χρειαζόταν ε, ε, μια συζήτηση. Φυσικά και δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφορετικότητα οικονομική. Προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε υποψηφίου από όλη την Ένωση. Παρ' όλα αυτά, εδώ βλέπετε μια πολύπλοκη εικόνα. Αλλά αν εστιάσετε στην τελευταία στήλη που λέει ποιοι έχουν προσληφθεί, στα δεξιά δηλαδή, Όσο πιο, χλωμό, όσο πιο αχνό είναι το χρώμα, τόσο πιο καλή είναι η ε, γεωγραφική κάλυψη. Μετά το 2010 αυτό αφορά 80% το 80% των διαγωνισμών. Το blue, μπλε το σκούρο έχουμε υπερπροσώπηση και το πράσινο δείχνει υπερπροσώπηση. Πολύ λίγα χρώματα σκούρα βλέπουμε και για προφανείς λόγους. Η Κροατία, χώρα προσχώρησης, το Βέλγιο, χώρα υποδοχής, ε, η Μάλτα που είναι το πιο μικρό ε, πληθυσμιακά κράτος μέλος ε, και γι' αυτό χρειάζεται τις ανάλογα πολλούς ε, γλωσσομαθείς να προσλάβουμε. Και κάτω-κάτω βέβαια, δεν σας εξηγώ, το Ηνωμένο Βασίλειο ουραγός. Και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα είναι πολύ πιο ισορροπημένη γιατί έχουμε πολύ πιο πολλά αχνά χρώματα. Αλλά δεν μας αρκούσε αυτό. Θελήσαμε να πάμε ακόμα πιο πέρα από αυτά που ήθελε το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, κάτι πολύ σημαντικό είναι. Δεν αρκεί να έχει μια καλή διαδικασία επιλογή. Πρέπει να προσελκύσει και του κατάλληλου υποψηφίου, να είσαι ελκυστικό εργοδότη. Θέλησαμε λοιπόν να λουστράρουμε την ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να, να, μπορεί να προσελκύει. Το 2009-2010 μηδέν ε, ήταν η αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών. Το 2016 το brand recognition αυτό είναι 15 ε, στον κατάλογο. Στο βαρόμετρο, το μεγαλύτερο βαρόμετρο του τέτοιου τύπου. Και στο δημόσιο τομέα στην πρώτη θέση είμαστε στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Που σημαίνει ότι όταν ε, οι τόποι υποψήφοι σκέφτονται το μέλλον τους, όλο και περισσότερο σκέφτονται μια καριέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και δεν περιμένουμε τους υποψηφίους να έρθουν σε εμάς, τους συνήθεις υπόπτους δηλαδή, αλλά εμείς τίνουμε ε, χείρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε 100 career ambassadors ε, ε, στην Ευρώπη και staff ambassadors που online ενημερώνουν τους δυνητικούς υποψηφίους. Τέλος, μας ασκήθηκε η κριτική το ότι δεν έχουμε αρκετές ε, πληροφορίες για τη διαχείριση, για τη διαχείριση και δεν είναι αξιόπιστα αυτές τις πληροφορίες. Σε σωστή και αυτή η κριτική. Τώρα έχουμε τα KPIs για τα περισσότερα από ό,τι κάνουμε, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Επίσης, κάτι άλλο που μας ε, ενδιαφέρει και είναι κάτι πολύ σημαντικό για την δική σας επιτροπή, είναι το κόστος. Και είχαμε μια εξαιρετική ε, μελέτη για το κόστος πρόσληψης ανθρώπων για το διεθνή δημόσιο τομέα. Δηλαδή είδαμε Παγκόσμια Τράπεζα, Εθνικό Ταμείο ή κτλ. Τότε ήμασταν ε, προς τα κάτω, από του πιο φθηνού, όπω βλέπετε στην δεξιά στήλη, σε σχέση με το μέσο όρο, που είναι πάνω από 40.000, ε, αν βάλουμε το σύνολο των δημόσιων, των εθνών οργανισμών. Προσπαθήσαμε με διοργανική συνεργασία το κόστος να μειωθεί κατά 1 τρίτο, ε, το ελέγχουμε και κάνουμε και κάποιες αλλαγές ανάλογα με το τι ε, θέση έχει προγεθεί αν είναι ASD e ή αν είναι AD. E και βλέπετε τις τιμές. Το κόστος ε, δεν έχει αυξηθεί όμως σε πραγματικούς όρους. Οπότε να συγκρίνεται με το κόστος πλήρους απασχόλησης, όχι μόνο στο λογικό κόστος. Και με βάση μια σταδιοδρομή 35 ετών. Λίγοι όπου να είναι δεύτερη θητεία μου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σας πω ποιες προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Που είναι και σοβαρές για όλα τα θεσμικά όργανα. Πρώτα απ' όλα γύρανση του πληθυσμού. Η γενιά των baby boomers απαχωρεί το 1 τρίτο του προσωπικού. Το 1 τρίτο στην Κομισιόν και το μισό του Κοινοβουλίου προσωπικό θα παρετηθεί. Θα, μάλλον θα αποσυρθεί λόγω σύνταξης. Επίσης είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσει ε, πολλοί δεν ενδιαφέρονται ούτε για να είναι πάντα στον ιδιοργοδότη, ούτε για να έχουν την ίδια καριέρα πάντα. Επίση θέλουν τελικά διαφορετικά είναι και πολύ διαφορετική οι σημερινοί υποψήφοι και θέλουν μια εργασία που να έχει νόημα. Αυτό είναι σημαντικό για τα θεσμικά όργανα. Εμεί έχουμε του προσφέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Το να έρθουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεισφέρουν στο μέλλον τη Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα, ε, ε, σταδιοδρομία, προαγωγές, πώς εργαζόμαστε, θεσμικά όργανα, τις τεχνολογίες κτλ. Αυτά δεν τους πολύ ελκύουν από ό,τι φαίνεται. Αυτό που βλέπουμε ε, όλο και περισσότερο και σε πολλές χώρες υπάρχει ανταγωνισμός προσέλκυσης ε, των πιο ταλαντούχων. Έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα ε, απασχόλησης ιστορικά και είναι δύσκολο να προσελκύσουμε άλλους. Υπάρχει επίσης και μια προσδοκία για το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να καθρεπτεί την διαφορετικότητα και την πολυμορφία. Το μέλλον άλλωστε ε, εξελίσσεται ε, πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να υπάρχουν ε, προφίλ διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια για να ολοκληρώσω. Πολλά ακόμα μπορούν να βελτιωθούν, πολλά έχουμε να κάνουμε. Καταφέραμε πάντως εμείς να καθιερωθούμε ως ένα κέντρο αριστείας στον τομέα μας και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερόμενους από όλα τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι μπορούμε να προσελκύσουμε ε, τους υποψηφίους. Επίσης μπορούμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές ε, με άλλα γραφεία οργάνωσης διαγωνισμών. Έχουμε αναγνωριστεί Υπήρξε και ένας γύρος τραπέζης ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ για τις καινοτομίες και τις βέλτιστες πρακτικές, στο οποίο συμμετείχαμε. Και στις τέσσερις πρώτες θέσεις, ε, τρεις, τέσσερις τώρα ήταν το 2015. Και έχουμε κερδίσει και πολλά άλλα βραβεία. Ελπίζω λοιπόν να βλέπετε ότι έχουμε πάρει πολύ σοβαρά υπόψη μας και αυτό που είπε το ελεγκτικό σύνδερο αλλά και όλες τις άλλες επικρίσεις που ακούστηκαν και σε ένα βαθμό ήταν δίκαιες. Και νομίζω ότι αρθήκαμε στο ύψος ε, των προκλήσεων. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πλέον προσφέρουμε πολύ καλύτερη υπηρεσία στους ε, θεσμούς ε, και δίνουμε ένα καλύτερο πρόσωπο θεσμών στους πολίτες που η μόνη επαφή είναι η έψω για να έρθουν κοντά στα θεσμικά όργανα. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν με δίκαιο τρόπο ή θα περάσουν ή δεν περάσουν. Ε, Εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε, να εξελισσόμαστε, να αλλάζουμε διαδικασίε. Μπορούμε και με την εμπειρία των υποψηφίων να βελτιωθούμε, να μειώσουμε και το χρόνο. Γιατί σε σχέση βέβαια ανάλογα και με τον κάθε κάστο του διαγωνισμού έχει δουλειά ακόμη το πράγμα. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρος. Πρέπει να σα πω ότι με εντυπωσιάσατε. Η κυρία Γιάλα Σέντε, έτσι το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή, η οποία απαντά στις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου στην ειδική του έκθεση του 2009. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ένθερμα τον κύριο Μπένφελτ ο οποίος ε, ουσιαστικά έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και έχει μεταμορφωθεί ε, σε έναν ε, μοντέρνο φορέα πρόσληψης υπηρεσία του. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν έχετε εντοπίσει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τα διάφορα θεσμικά όργανα. Αν μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν κάποια κέντρα που είναι πιο ελκυστικά ή όχι, ανάλογα με το πώς παρουσιάζονται, η ΕΝΙΕΦΣΟ ε, κάνει μία ομοιόμορφη παρουσίαση όλων των κέντρων. Θα ήθελα να μου πείτε δηλαδή αν ε, φτάνουν ε, από κάποια θεσμικά όργανα ε, κάποια πιο, κάποια πιο μορφότυπη για την πρόσληψη. Επίσης, να μας πείτε ποια είναι η σχέση σας με ανθρώπους που έρχονται και κάνουν μια πρακτική, παραδείγματος χάρη, από τις ε, εθνικές δικήσεις ε, και με ανθρώπους που έχουν πάρει υποτροφίες. Εσείς ε, μπορείτε να μας πείτε και αν έχετε κάποια αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή αν τελικά οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται βελτιώνονται για να μπορούν στη συνέχεια να περάσουν τις εξετάσεις. Λοιπόν, επίσης θέλω να μου πείτε αν έχουμε δει τον αντίκτυπο της κρίσης, ε, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση της ε, χώρας μου, Σίγουρα οι θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει μια πόρτα εξόδου για νέους που δεν έβρισκαν δουλειά στην Ισπανία. Έχει γίνει κάτι τέτοιο ισχύ και για τις υπόλοιπες εθνικότητες. Και επίσης, όπως ε, είδαμε, το θέμα του μισθού μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό, όμως ε, στην ε, περίπτωση ορισμένων κρατών μελών, μπορεί, παίρνοντα χάρη, να παίζει ρόλο και το θέμα του μισθού, αν υπάρχει υποβάθμιση του επίπεδου ζωή. Υπάρχει και κάτι άλλο που μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Έχετε κάποια φόρμουλα για να μετρήσετε την ε, δεύτερη ή τρίτη γενιά υπαλλήλων που έρχονται από άλλε χώρε. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μια ανοιχτή πόρτα για να μπουν άτομα που έχουν άλλο background. Όχι καθαρά το ευρωπαϊκό, δηλαδή μπορεί να έρχονται παραδείγματο χάρη από οικογένειε μεταναστών. Ίσως ε, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα που έχουμε, καθώς ε, έχουμε γύρωση του πληθυσμού. Παρακαλώ, κύριε Σιλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της ΕΠΣ για την παρουσίασή του. Σίγουρα η διαχείριση της επιλογής προσωπικού είναι μια πολύ πολύπλοκη δραστηριότητα. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το ένα το παρουσίασε η κυρία Γιάλα, αλλά εγώ θα το πω από μια άλλη οπτική. Να ρωτήσω αν ε, η κρίση, όχι η οικονομική κρίση, αλλά η κρίση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ε, έχει κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει τον αριθμό των νέων ε, που θέλουν να εργαστούν σε θεσμικά όργανα, δηλαδή τη δέσμευσή τους με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αφενός και δεύτερον τους λόγους ασφάλειας Παίρνουμε χάρη η ασφάλεια που παρουσιάζεται να μπουν ε, ω εργαζόμενοι στα θεσμικά όργανα ε, Βλέπετε δηλαδή έλλειμμα ενδιαφέροντος ή αντιθέτως ε, υπάρχει ζήτηση, έχει διατηρηθεί ζήτηση. Επίσης μιλήσαμε τώρα για το θέμα το γενολογικό, ένα μεγάλο μέρος των υπαλλήλων θα συνταξιωτηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς λειτουργεί το σύστημα της πρόληψης πριν οι διαδικασίες επιλογής ήταν πιο προσανατολισμένες στο θέμα του προσανατολισμού και της εμπειρίας. Και θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε να κάνετε μια αξιολόγηση των διαδικασιών επιλογής. Και μια τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε. Πολλές φορές η κατάρτιση ε, καταλόγων ε, καταλόγων των επιτυχόντων ε, σημαίνει ότι ε, κάποιος δεν θα έχει σίγουρη ε, θέση. Πώς ε, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη δόση διαφάνειας για να υποστηρίξουμε τους πλέον ικανούς που μπαίνουν σε αυτούς τους καταλόγους. Um Κύριε Κάντεμπαχ, πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Δεν εντασσόταν στις συστάσεις βέβαια του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξέρουμε τι πιστεύετε σε σχέση με τις πρακτικές, διότι στη διαδικασία αυτή προσλήψεων βοηθάει αν ε, υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε περιόδους άσκησης ε, πρακτικής ε, γιατί αποκτούν εμπειρία. Το έχουμε δει και σε διαδικασίες διαγωνισμών ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποιοι ατυπικοί σταζιέρ κατά κάποιο τρόπο που δεν ξέρουν ακριβώς πώς πάει η διαδικασία, δεν υπάρχει διαφάνεια. Εσείς ε, έχετε να κάνετε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο μέλλον και ο κ. Λιμπεράτσκι σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Βλέπουμε ότι γίνονται αλλαγές προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας πρόσληψης. Πολύ συχνά Ακούω παράπονα ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η διαδικασία, ότι δεν είναι διαφανής, δεν είναι σαφής. Και τονίζονται κάποια θέματα όπως το θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας. Αν πάρουμε δύο χώρες συγκρίσιμες σε μέγεθος, την Ισπανία και την Πολωνία, από την πολωνική πλευρά έχουμε τρεις φορές λιγότερες αιτήσει από την Ισπανία όμως και πέντε φορές ε, λιγότερο επιλεγμένα άτομα. Έτσι λοιπόν έχουμε υπερεκπροσώπηση της Ισπανίας που δεν είναι και τόσο μεγάλη και δεν θα έπρεπε να παραπονιέται τόσο πολύ. Όμως σίγουρα μια χώρα όπως η Πολωνία υποεκπροσωπείται. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι προτιμούνται κάποιοι υποψήφοι από συγκεκριμένε χώρε. Ποια είναι η αιτία, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα του συγκεκριμένου κράτου μέλου ή το μοντέλο σταδιοδρομία ή κάτι άλλο. Και η επόμενη ερώτηση. Έχουμε κάποια ανάλυση της ε, επάρκειας ε, της ίδιας της διαδικασίας ε, επιλογής, δηλαδή αν έχει γίνει σωστή η επιλογή του προσωπικού και ήταν ορθή ή όχι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παρακαλώ σύντομα να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Προφανώς η ΕΠΣΟ απαντώντας στην πρώτη ερώτηση, επιδιώκει να προσλάβει ανθρώπους με, για όλα τα θεσμικά όργανα και συζητάμε για τους ρόλ, διαφορετικούς ρόλους των θεσμικών οργάνων και την τοποθεσία τους. Σαφώς κάποια θεσμικά όργανα έχουν, είναι πιο προβεβλημένα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ άλλα είναι λιγότερα ελκυστικά. Αλλά παρόλα αυτά ε, προσλαμβάνουν αυτούς που χρειάζονται. Υπάρχει και κάποια διαφορετική, διαφορετική ελκυστικότητα ε, γεωγραφικά. Είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσουμε προσελκύσει κανεί ανθρώπου για το Λουξεμβούργο πρώτη για τι Βρυξέλλες για διάφορους λόγου, ενδεχομένω το κόστο ζωή είναι ένα βασικό παράγων στην περίπτωση αυτή. Η ΕΠΣΟ δεν ε, παίζει ρόλο όσον αφορά την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων, αυτό είναι θέμα των θεσμικών οργάνων, δεν μπορώ να πω τίποτα. Όσον αφορά τους ε, σταζιέρ, τους εκπαιδευόμενους, ε, αυτούς που είναι σε μαθητεία. Είναι ένα σημαντικό μια σημαντική δεξαμενή ταλέντου για τα θεσμικά όργανα και συνεργαζόμαστε με τα διάφορα έργα μαθητείας των θεσμικών οργάνων για να συναντούμε τα άτομα αυτά στη διάρκεια της μαθητείας τους. Τους εξηγούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για διαδρομία, πώς μπορούν να γίνουν ε, να κάνουν αίτηση πρόσληψης και πολλοί από αυτούς οι οποίοι προσλαμβάνονται ε, είναι άτομα που έχουν περάσει από μαθητεία. Δηλαδή βλέπουμε την ε, πορεία αυτών των ανθρώπων που ξεκινάνε από μαθητεία, μετά έχουν κάποια σύμβαση και στο τέλος γίνονται υπάλληλοι. Είναι άτομα με μεγάλο ταλέντο που έχουν δείξει ήδη ότι ενδιαφέρονται να εργαστούν για, την, ε, για τα θεσμικά όργανα. Βεβαίως η οικονομική κρίση είχε επηρέασε τη δουλειά μας, σαφώς. Ακόμα και τόσα χρόνια εργότερα. Το γεγονό ότι υπάρχει τόσο ψηλό ποσοστό ανεργία νέων σε πολλά κρατημέλη, κυρίω στην Νότια Ευρώπη, έχει ε, δώσει αυξημένου αριθμού αιτήσεων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, όπω ήταν αναμενόμενο. Και εξίσου βλέπει κανεί ότι σε χώρε όπου η Γερμανία, που υπάρχει υψηλό επίπεδο απασχόληση, υψηλό επίπεδο ζωή, ε, υψηλό επίπεδο ε, στοιχειούχων δύσκολα προσλαμβάνει κανείς από εκεί. Ο, ο, ο μισθός παίζει ρόλο, είναι ελκυστικό να εργάζεται κανείς εδώ όταν ε, προέρχεται από κανείς από κράτη μέλος που ο βασικός μισθός είναι εκατοντάδες και χιλιάδες. Αλλά αν θέλουμε να προσελκύσουμε άτομα από την Δανία είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουμε. Η μισθή είναι υψηλή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που υπησέρχονται όπως η στάση απέναντι στην Ευρώπη, η ποιότητα, θέματα ποιότητα ζωής. Σε ε, υπάρχουν χώρε που εν γέννη ποιότητα ζωής είναι πολύ ψηλή και δεν έχει αυτό σχέση μόνο με τα χρήματα. Πρόσφατα ακούσαμε από διάφορα κράτη-μέλη ότι οι Βρυξέλλες απο, αποδεικνύεται πρόβλημα μετά τις τρομοκρατικέ επιθέσεις που έγιναν πέρσι. Πολλοί το ξανασκέφτονται για το να έρθουν στις Βρυξέλλες, δικαίω ή αδίκω, αλλά πάντως επισέρχεται αυτό το θέμα. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στην πολυμορφία και έχουμε μελετήσει τις ροές ε, ανθρώπων λεπτομερώς που ε, με βάση από τους, του διαγωνισμού του 85 και ε, προέρχονται από διαφορετική διαφορετικούς κλάδους, διαφορετικά πανεπιστήμια και υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πολυμορφία, όχι όμως επαρκή. Υπάρχει, από, υπάρχουν υποψήφοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για τους μετανάστες πρέπει να έχουν διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πέραν αυτού δεν υπάρχει ε, άλλο εμπόδιο. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία, υποψήφιους με αναπηρία. Αυτό ε, απαιτεί προσπάθεια και από τα θεσμικά όργανα φυσικά. Δεν βλέπουμε... Ε, κάποια κρίση να δημιουργείται, κρίση εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Αντίθετα, μεταξύ των νέων θεωρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον που προκαλείται και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Θεωρούν ότι είναι μια ε, εξαιρετική ευκαιρία για αυτούς να συνεισφέρουν, να προσφέρουν στην κοινωνία. Είναι ε, αντίθετο από αυτό που θα περίμενε κανείς, αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Θεωρούμε ότι η τα κίνητρα δεν μετρώνται από τις, πολλές, τις παλαιές, ε, τα πολλά τεστ, πολλά επιλογής που ήταν αδύνατο να τα περάσει κανείς. Αν δεν ζούσε στις Βρυξέλλες δεν είχε πρόσβαση στα βιβλία με τις 250 ερωτήσεις κτλ. Αλλά ε, ε, ελέγχουμε τις γνώσεις αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο για να καταλάβουμε ότι υπάρχει κατανόηση και αν υπάρχει κίνητρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Προσπαθούμε να ελέγξουμε τα κίνητρα των ανθρώπων όταν έρχονται εδώ και θεωρούμε ότι αυτοί που έρχονται έχουν κίνητρο. Και έχει γίνει για πολλά χρόνια μια μελέτη στην Κομισιόν και δεν υπάρχει ε, πτώση των κινήτρων ε, δεν, οι άνθρωποι έχουν την ίδια κινητοποίηση όπως και πριν από 10 χρόνια. Όσον αφορά τον κατάλογο εναν, αυτών που είναι εν αναμονή έχουμε βελτιώσει πολύ. Οι πιθανότητες πλέον να προσληφθεί κανείς είναι πολύ ψηλότερες. Όλες οι θέσεις για τους επιτυχόντες είναι ε, δημοσιευμένες. Προηγουμένως έπρεπε κάποιον να ξέρεις, να ψάξει και να σου πει πού να πας αυτό είναι άδικο θα έλεγα, βασικά άδικο. Τα πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ίσως θα πρέπει να ε, είναι διατεθειμένα τα θεσμικά όργανα να κλείσουν κάποιου από του παλιού καταλόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά πάει το πράγμα. Όσον αφορά το θέμα των, ε, αυτών που είναι σε μαθητεία, το ανέφερα αυτό. Υπάρχει ένα ταλέντο εκεί, μια δεξαμενή ταλέντων. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε μόνο επιπληρωμή ε, άτομα σε μαθητεία, αλλά συνεργαζόμαστε πολύ στενά μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό που βλέπουμε σε άλλους οργανισμούς παγκοσμίως υπάρχει μια πιο ε, στενή σχέση μεταξύ της μαθητείας και της χρήσης ως δεξαμενή ταλέντου. Δηλαδή έχει κανείς τη δυνατότητα και μετά μέσα από ένα διαφορετικό δρόμο περνάει στην απασχόληση. Ενώ εδώ υπάρχει μια τελεία όταν τελειώσει η μαθητεία και μετά πρέπει κανείς να ξαναρχίσει. Είναι θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα. Ξεπερνά τη δική μας, το δικό μας πεδίο αρμοδιότητες. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που περνούν τους διαγωνισμούς που ο προηγούμενος ε, εργοδότης τους ήταν κάποιο θεσμικό όργανο της Ένωσης. Δηλαδή προσελκύουμε άτομα για κάποιο διάστημα και σαφώς ανακαλύπτουν ότι ενδιαφέρονται να δουλέψουν για την Ευρώπη και θέλουν να παραμείνουν. Τέλος, Θεωρώ ότι είμαστε εξαιρετικά διαφανείς σε κάθε φάση της διαδικασίας επιλογής. Δημοσιεύουμε πληροφορίες για όλους. Όλοι ενημερώνονται για τους βαθμούς τους. Όποιος έρχεται στο κέντρο ε, αξιολόγησης, είτε περάσουν είτε δεν περάσουν, έχουν, ε, παραλαμβάνουν μια αναφορά με παρατηρήσεις, όχι μόνο τους βαθμούς τους, για το πώς πήγαν, είτε πέτυχαν είτε απέτυχαν. Νομίζω ότι σαφώς υπάρχει ένα θέμα ε, για τους υποψηφίους από κάποια κράτη-μέλη. Έχουμε ε, πρόβλημα να προσελκύσουμε τους κατάλληλους ε, υποψηφίους από την Πολωνία. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Το μελετάμε με τις αρχές. Έχουμε κάνει, οργανώσει ένα σεμινάριο το φθινόπωρο με, για τις χώρες, από τις 7 χώρες που είναι δύσκολο να προσελκύσουμε ανθρώπους και ε, θα καλέσουμε εκπροσώπους από την ε, πολωνική κυβέρνηση. Θέλουμε να καταλάβουμε ποια είναι η ιδιαιτερότητα κάθε κράτους μέλους για να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε το σωστό για να προσελκύσουμε τους σωστούς σε σενή συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις για να γνωρίσουν, γιατί εκείνες γνωρίζουν την κατάσταση επιτόπου καλύτερα από εμά. Να κάνουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους για κάθε κράτος μέλος στους, στα θεσμικά μας όργανα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με έχει εντυπωσιάσει η συνέχεια που δώσατε σε αυτές τις συστάσεις. Σίγουρα πρέπει να συνεχίσετε στον καλό αυτό δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν η ΕΠΣΟ να δείχνει ότι συνεχίζει να προσπαθεί να εφαρμόσει τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου.